Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ας ε, περάσουμε στην Task Force Τουρισμού της Επιτροπής μας. Η κυρία Τέλη μου ζήτησε να προεδρεύσω εγώ σήμερα στην ομάδα αυτή. Γι' αυτό και βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους όσοι ήρθατε από τις διάφορες οργανώσεις τουρισμού, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου έχουμε μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα. Και αργότερα θα έχουμε και ένα σημαντικό στέλεχος του ΟΗΕ για τον τουρισμό. Θα μιλήσουμε περισσότερο για το έτος τουρισμού Κίνα Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω το λόγο ε, στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Grow. Ο κύριος Μερτομάκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα θέματα του τουρισμού και σίγουρα θα υπάρχουν μετά και ευρωβουλευτές που θα θέλουν να πάρουν το λόγο. Οπότε, Γενική Διεύθυνση Γκρό, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μας να μπορέσουμε να σας πούμε Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το έτος τουρισμού 2018 Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα. Είμαστε στο πρώτο στάδιο της υλοποίησης, πάντως ήρθα εδώ για να σας ενημερώσω πώς θα προχωρήσει η υλοποίηση αυτή. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τους οικονομικούς δεσμούς ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα. Η Κίνα είναι ο πρώτος εταίρος όσον αφορά τις εισαγωγές, αλλά και τις εξαγωγές νομίζω για μας η Κίνα έρχεται στη δεύτερη θέση. Οι σχέσεις μας έχουν ενισχυθεί. Και γι' αυτό θελήσαμε να ασχοληθούμε και με αυτή την ανθρώπινη διάσταση. Ο πρόεδρος ε, Γιούνκερ λοιπόν αποφάσισε να ξεκινήσει το 2018 ως έτος τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Να σας πω ποια είναι τα κύρια στοιχεία που βλέπουμε. Υπάρχουν διμερείς σχέσεις βέβαια αλλά στους στόχους μας θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα θέλουμε να ενισχύσουμε την αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στους Ευρωπαίους και τους Κινέζους, η ανθρώπινη διάσταση δηλαδή. Δεύτερον, θέλουμε περισσότεροι Κινέζοι να έρχονται και να επισκέπτονται τα μέρη μας και να μαθαίνουν ε, την οτροπία μας, τον πολιτισμό μας. Άρα πάλι είναι ανθρώπινη διάσταση εδώ και βέβαια να υπάρξουν και περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κίνα. Αυτή είναι η οικονομική διάσταση. Από τη δικιά μας την πλευρά μπορώ να σας πω ότι έχουμε κάποιους ειδικούς στόχους. Θέλουμε να προωθήσουμε το βιώσιμο τουρισμό θέλουμε οι Κινέζοι να πάνε και σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς και όχι σε αυτούς που συνέχεια επισκέπτονται. Έτσι πιστεύουμε θα ενισχύσουμε την ανάπτυξη και θα την μοιράσουμε σε ολόκληρη την επικράτεια. Έπειτα θέλουμε να ενισχύσουμε τις επενδυτικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας. Θα πρέπει να μην υπάρχουν πια φραγμοί στις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην Κίνα και νομίζω ότι ε, τώρα θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις γι' αυτό. Έχοντας όλα αυτά υπόψη μέσα στη χρονιά, θα προχωρήσουμε σε διάφορες δραστηριότητες. Πρώτα απ' όλα θα βοηθήσουμε τους τουριστικούς παράγοντες, φορείς, ε, ε, τουριστικές οργανώσεις, επιχειρήσεις κλπ. με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Πρέπει να πάτε στην ιστοσελίδα μας του έτους τουρισμού 2018 Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα και εκεί θα βρείτε πολλά στοιχεία. Επίσης θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες τουριστικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας με τους Κινέζους εταίρους. Οργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις μεταξύ επιχειρήσεων υπέρ του τουρισμού και η δουλειά έχει προετοιμαστεί ε, με το πειραματικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον τουρισμό με την Κίνα. Σε πολλές ε, τέτοιες εκδηλώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, ο προσκεκλημένος, ο προσκεκλημένος και είναι κάτι που θα συνεχιστεί μέχρι και τον Αύριο. Και τρίτον προχωρούμε ώστε να προωθήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά. Εξού και έχουμε προωθήσει μια νέα πρωτοβουλία, μια πλατφόρμα, κάτι το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα νέο εργαλείο έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν δράσεις που προωθούν την Ευρώπη στην Κίνα και θα μας βοηθήσει να μάθουν οι Κινέζοι περισσότερα για τον τουρισμό στις χώρες μας, για την πολιτιστική μας κληρονομιά, για περισσότερους προορισμούς κλπ. Επίσης θέλουμε να οργανωθούν περισσότερες εκδηλώσεις ώστε να βρεθούν πιο κοντά οι Ευρωπαίοι με τους Κινέζους. Ήδη στην Grand Place, για παράδειγμα, είχαμε τα γένεια μιας τέτοιας πρωτοβουλίας στις 22 Φεβρουαρίου. 2 Μαρτίου τώρα διάφορα κτίρια θα φωτιστούν κόκκινο. Ε, κάτι το οποίο γίνεται προς τιμή του Κινέζικου Φεστιβάλ Φώτων. Όλες αυτές οι δραστηριότητες θέλουμε βέβαια να αποφέρουν καρπούς. Έχουμε βάλει κάποια στοιχεία. 200 νέες ε, συμφωνίες εταιρική σχέσης θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις με την Κίνα. Αύξηση επίσης κατά 10% των Κινέζων τουριστών σε σχέση με σήμερα και αυτό να συνεχιστεί κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ένα δισεκατομμύριο το χρόνο για την ευρωπαϊκή οικονομία, επιπλέον έσοδα δηλαδή. Και όλα αυτά θέλουμε να τα κάνουμε βέβαια σεβόμενοι τις ανάγκες των τομικών κοινωνιτήτων. Με βιώσιμο τρόπο δηλαδή. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι δουλεύουμε σκληρά για την υλοποίηση της εμβληματικής πρωτοβουλίας και για να πετύχουμε χρειαζόμαστε στενή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη, αλλά και με τις περιφέρειες και τους Δήμους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια. Έχει μεγάλη σημασία για την υλοποίηση του έτους τουρισμού Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τη φωνή της Κομισιόν. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τους συναδέλφους που θα ήθελαν να κάνουν ερωτήσεις ή να εκφράσουν τις απόψεις τους για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού να πάρουν το λόγο. Κλάουντια Μοντέρο Αγιλάρου και ο Βιμ Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω για την παρουσίαση σχετικά με αυτούς τους στόχους και τις προτεραιότητες που περιγράφησαν και που πρέπει να επεξεργαστούμε για να προωθήσουμε αυτό το έτος ευρωπαϊκού ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και ήθελα να τονίσω ότι είναι τέσσερα τα σημεία που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και θα ήθελα να ρωτήσω με τι μορφή θα οργανωθούν συγκεκριμένες δράσεις τι μορφή θα πάρουν δηλαδή συγκεκριμένες δράσεις. Η πρόθεση των βιώσιμων προορισμών, του βιώσιμου τουρισμού δηλαδή, με τι δράσεις θα επενδυθεί αυτή η βιωσιμότητα για να προωθήσουμε όλη την Ευρώπη προς τους Κινέζους, διατηρώντας όμως τα χαρακτηριστικά των τοπικών προϊόντων, των ιδιαίτερων υπηρεσιών που προσφέρει ο καθένας και μαζί κάποιες ιδιαιτερότητες κάποιων περιοχών της Ευρώπης. Πώς θα παρουσιαστεί αυτό, πώς θα εκφραστεί στην ε, μελλοντική δράση. Επίσης, ε, προφανώς συμφωνώ με την ανάγκη να διευκολυνθεί η έκδοση θεωρήσεων. Ξέρουμε ότι ως προς τις θεωρήσεις η κατάσταση έχει κάπως ε, μπλοκαριστεί στο κοινοβουλευτικό μας έργο, γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προβλέψει κάποιο άνοιγμα, έχοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που ληφθούν υπόψη, την ασφάλεια και όλες τις προκλήσεις που αυτή τη στιγμή βιώνουμε στην Ευρώπη, όμως ε, για την διευκόλυνση των ε, θεωρήσεων τι συμβαίνει ακριβώς με αυτό το συγκεκριμένο ε, σημείο. Και επιπλέον, για να ολοκληρώσω, σε αυτή την πρώτη παρέμβαση, προβλέπουμε αύξηση του αριθμού των επισκεπτών από την Κίνα. Συγκεκριμένα, πώς θα προωθηθεί η αύξηση των αφήξεων εδώ. κάποιες περιοχές ε, ε, της Ευρώπης θα πρέπει να λάβουν ιδιαίτερη μέρημνα ίσως. Προωθούμε λοιπόν συνολικά το προϊόν Ευρώπη ως τουριστικό προϊόν. Ποιες είναι οι ιδέες που βρίσκονται επιτάπτως. Σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την πρωτοβουλία, διότι πράγματι οι σχέσεις μας από παλιά είναι καλές σχέσεις και στην Πορτογαλία βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη θέση λόγω ιστορικής, ε, ιστορικών λόγων με την Κίνα. Υπάρχει λοιπόν, ε, υπάρχουν στενές σχέσεις λόγω της οικονομίας αλλά και η διασταύρωση πολιτιστική, η Συναντήσει οι πολιτιστικέ είναι σημαντικέ για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις σημερινές, προκλήσει τη κοινωνία προκλήσεις της κοινωνίας μας. Κοινωνίες που ζούμε και που θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε καλύτερη σύσφυξη των σχέσεων. Θα ήθελα λοιπόν να παραμείνω σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, Κλάουντια. Θα δώσω το λόγο σε μένα τον ίδιο, όσο προβλεφτεί και θα μιλήσω ουγγρικά. Ίσως και να με καταλάβετε. Ή χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας. Συνάδελφοι, η πρόταση συναδελφοι αυτη την πρόταση αυτή την έκανα από τριετίας, να έχουμε ένα θεματικό έτος τουρισμού Ευρώπης-Κίνας. Και νομίζω ότι έχουμε επαναπαυθεί στις δάφνες μας εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε χάσει την αρχική ορμή που θα μπορούσαμε να είχαμε σε αυτή την πρωτοβουλία. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η συνεργασία με την Κίνα σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα είναι ε, ύψης της σημασίας για την Ευρώπη. Αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος Τουρισμού Ευρώπης-Κίνας είναι 365 μέρες, ε, μια σειρά από εκδηλώσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, ε, συναντήσεις διεπιχειρησιακές. Όμως σίγουρα δεν θα αλλάξουμε μέσα σε μια χρονιά ε, τον κόσμο και τις ευρωκινέζικες σχέσεις με την διοργάνωση ενός τέτοιου έτους. Το ερώτημα λοιπόν είναι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το έτος για να επικεντρωθούμε σωστά στο θέμα, στον τομέα του τουρισμού. Θα μπορέσουν οι πολιτικοί και οι θύνοντες, όσοι λαμβάνουν αποφάσεις, να αρχίσουν να σκέφτονται με κινέζικούς όρους, να υιοθετήσουν τον κινέζικο τρόπο σκέψης. Ε, χάρη στους ε, διοργανωτές αυτής της ημερίδας και τον κύριο Σανταντέρ, ε, ήδη προς τα τέλη Φεβρουαρίου βλέπουμε ότι το έτος ε, τουρισμού Ευρώπης-Κίνας αρχίζει να προβάλλεται παντού. Βλέπουμε λοιπόν φως στην άκρη του τούνελ και όχι μόνο χάρη στην ανακτήρια τελετή, αλλά χάρη στο γεγονός ότι όλα και περισσότερα κράτη-μέλη και οργανώσεις τους αρχίζουν να παίρνουν σοβαρά το όλο θέμα. Θέλουν να έχουν εμπορικές σχέσεις με την Κίνα. στατιστικά στοιχεία πρόσφατα έχετε δει, διότι εάν δεν τα γνωρίζετε, να σας δώσω εγώ κάποια. Ε, πολύ πρόσφατα είχαμε μία εβδομάδα διακοπές ε, στην Κίνα λόγω πρωτοχρονιάς. Η χρονιά του σκύλου ε, ξεκίνησε πρόσφατα. Και έφυγε μεγάλος αριθμός τουριστών από τη χώρα ανάλογος με αυτόν των τουριστών που φεύγουν από την Ευρώπη μέσα σε ένα ολόκληρο χρόνο. Μιλάμε για πολύ κόσμο, πολλοί Κινέζοι τουρίστες. Και αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος της μέσης τάξης των Κινέζων που έρχονται καθημερινά στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν κάπως πρέπει να το σκεφτούμε. Εδώ, σε αυτό το δωμάτιο, σε αυτή την ομάδα δράσης, έχουμε ασχοληθεί με το θέμα του τουρισμού. Αν ρωτήσετε τον κόσμο που ζει στην Βαρκελόνη, στη Βενετία ας πούμε, θέλετε έξι φορές παραπάνω Κινέζους τουρίστες ε, στο πικ της ε, τουριστικής σεζόν, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Μπορεί και να πούνε όχι, αλλά δεν θα πάρουμε. Δεν μπορούμε να τους ε, βολέψουμε τόσους πολλούς. Θα πρέπει λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να αρχίσουν να σκέφτονται Πώς μπορούμε από τις Βρυξέλλες, από το ευρωπαϊκό επίπεδο να βοηθήσουμε, να διευκολύνουμε τους τοπικούς φορείς του τουρισμού, ώστε να ωφεληθούν από την έλευση τόσων πολλών Κινέζων. Η εποχικότητα λόγω χάρη είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Πώς μπορούμε να προσελκύσουμε και να στεγάσουμε, να ε, φροντίσουμε για την ε, στέγαση τόσων Κινέζων τουριστών. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται σε όλη την περίοδο της τουριστικής σεζόν, ε, όχι μόνο στι περίοδου αιχμής. Να φροντίσουμε να υπάρξει επέκταση αυτών των ε, περίοδων. Πηγαίνω συχνά στην Κίνα και έχω συχνά συνομιλίε με υπευθύνου του τουριστικού κλάδου Και πολλέ φορέ ε, και αυτοί οι ίδιοι δεν γνωρίζουν σημαντικού ευρωπαϊκού προορισμού. Ξέρουν 5-6 βασικού προορισμού και όλοι θέλουν να πάνε σε αυτού του 5-6, 8-10 βασικού προορισμού. Βεβαίω, δεν μπορούμε να περιμένουμε οι ισπανικέ ή οι ιταλικές αρχές, οι οργανισμοί τουρισμού τη κάθε χώρα να του πούν πηγαίνετε στην Πράγα ή στη Βουδαπέστη να την έρθετε σε εμά ή γιατί δεν πάτε στη Φιλανδία, ένα πολύ όμορφη χώρα. Προφανώ του θέλουν. Οι τοπικέ αρχέ ε, κοιτάζουν να εξυπηρετήσουν τα τοπικά συμφέροντα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε τον τρόπο σκέψη μα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να σκεφτούμε τι εκστρατείε διαφήμιση, πρόθεση μπορούμε να οργανώσουμε. Μια ε, σφαιρική στρατηγική ε, στην Ευρώπη που να καλύπτει ολόκληρο το μεριολογιακό έτο και όλε τι ευρωπαϊκέ περιοχέ. και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πιο ε, ισότιμη κατανομή και γεωγραφική και ημερολογική. Οι εθνικοί οργανισμοί τουρισμού. Εμείς ε, στο Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει από κοινού να αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Είναι δική μας ευθύνη. Δεν θέλω όμως να μακρηγορήσω, ούτε να μονοπολίσω το χρόνο αγόρευσης. Και σας καλώ όλους, όπως έκανα και γραπτός, σας καλώ όλους στην αυριανή μεγάλη διάσκεψη που είναι μια από τις βασικές εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Έτους ε, Τουρισμού Ευρώπης-Κίνας. Θα κηρύξει την έναρξη ο πρόεδρος Ταγιάννη. Θα υπάρξουν εκατοντάδες συμμετέχοντες, Κινέζοι και Ευρωπαίοι, θύνοντες, ε, φορείς, και οι μεγαλύτεροι οργανισμοί της Ευρώπης. Οργανισμοί τουρισμού. Σας προσκαλώ λοιπόν εφόσον θέλετε να ξέρετε περισσότερα για αυτό το θέμα. αυτά είχα να πω ως Προεδρεύων και Ε, αυτή η μισάωρη συζήτηση που οργανώσαμε εδώ σε αυτή την αίθουσα δεν σημαίνει ότι έκλεισε το θέμα. Θα ξανασχοληθούμε με αυτό πριν λήξει το Ευρωπαϊκό Έτος Τουρισμού Ευρώπης Κίνας και να δούμε τι μπορεί να γίνει και σε άλλα επίπεδα. Θα μας απασχολήσει ας πούμε αν μπορούμε μελλοντικά να οργανώσουμε κάτι ανάλογο και για τον τουρισμό των Ινδών Θέλουμε να καλωσορίσουμε Κινέζους τουρίστες στην Ευρώπη και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για την Κίνα, την ε, κινέζικη νοοτροπία και τον κινέζικο πολιτισμό και πώς και οι Ευρωπαίοι μπορούν να πάνε να επισκεφτούν την Κίνα. Να το έχουμε και αυτό κατά νου, ώστε αυτές οι σχέσεις να είναι περισσότερο ισότιμες. Ο κύριος Φάντενκάμπ έχει το λόγο. Έχετε σχόλια, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό σας για τις τουριστικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα. Εννοείται, είναι υπέροχο. Και ευχαριστώ και τον κύριο Πελτομάκη για την παρουσίασή του. Δύο ερωτήσεις έχω. Η Κλάουντια αναφέρθηκε ήδη στο θέμα των θεωρήσεων, των βίζα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω περισσότερα τι γίνεται με αυτό. Έχει λυθεί, έχει απλοποιηθεί το θέμα και επίση θέλω να ξέρω ποιες είναι οι συνέπειες από το Brexit. Υπάρχουν επίσης αρκετά ξενοδοχεία Υπάρχουν αρκετοί ξεναγοί που νομιλούν κινέζικα. Υπάρχουν ε, Υπάρχει αρκετό κινέζικο φαγητό, γιατί δεν νομίζω ότι θα τρώνε πατάτες τηγανιτές με μαγιονέζα. Αυτά τα πρακτικά θέλω να μάθω. Η μεσαία τάξη αυτή που είναι 700 εκατομμύρια Κινέζοι, ναι, καλύτερα να μην μας έρθουν όλοι μαζί, γιατί δεν θα μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε βέβαια. Όμω, να ξέρετε ότι συμμετέχω στην αντιπροσωπεία για τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Κίνα και στην αντιπροσωπεία αυτή, να ξέρετε, έχουμε μια βασική έννοια και αυτή είναι η έννοια της αμοιβαιότητας. Κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνεται πάντα η Κίνα, τουλάχιστον όχι με τον ίδιο τρόπο που τα λαμβανόμαστε εμείς στην Ευρώπη. Γι' αυτό η ερώτηση προς τον κύριο Πελτομάκη είναι οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες έχουν ε, τις ίδιες δυνατότητες να στείλουν ας πούμε τους δικούς μας ε, συνταξιούχους στην Κίνα με τους δικούς τους ε, ξεναγούς να βρίσκουν τα φαγητά που τρώνε εκεί κτλ. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα στις σχέσεις και είναι κάτι που δεν υπάρχει στη βιομηχανία όσον αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρωτάω κατά πόσο στον τουρισμό υπάρχει. Γιατί βέβαια και εγώ λαδό είμαι και εγώ θέλω να βγάλω λεφτά από την Κίνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τεγκράντης Πασκουάλ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ο συντονιστής μου, Βιν μου είπε, είπε τα βασικά ε, που με ανησυχούν. Πράγματι, η αμοιβαιότητα είναι ένα ζήτημα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί Η Η Realpolitik μας έχει κάνει να μην βλέπουμε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Κίνα. Έτσι έχει η πραγματικότητα. Και κάποιους ε, Αμερικάνος ζήτησε και βοήθεια από την Κίνα και μα δεν ξέρουν τι είναι η Wall Street. Δεν υπάρχει αμοιβαιότητα. Έρχονται κάποιοι για να εργαστούν, να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, είναι αποτελεσματικοί και ανοίγουν το μυαλό τους και τη ζωή τους και έπειτα είναι και οι πλούσιοι στα μεγάλα καταστήματα τα πιο πολυτελή έχουν Κινέζους ως ε, υπαλλήλους. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η οικονομική παρουσία των πλούσιων Κινέζων. Αυτή είναι πραγματικότητα. Αν έρχονται όλοι, όχι, δεν έρχονται όλοι. Είχα πάει στην Κίνα με άλλη ιδιότητα, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και τότε το μήνυμα ήταν πρώτοι θα περιμένουν, μάλλον πρώτοι θα δουν την ευημερία στην Κίνα και τον εξυγχρονισμό και οι υπόλοιποι θα περιμένουν. 40.000 δημοσιογράφοι ε, βλέπουν ότι, άλλοι, ότι στην Κίνα απλά δεν κυκλοφορούν με ποδήλατα αλλά με Audi. Ιντερνετ. Και είδαμε τι και με το ίντερνετ που είναι η άλλη πλευρά. Πρέπει λοιπόν να δούμε την πραγματικότητα. Εμείς πρέπει να σεβαστούμε βέβαια τα θεμητά συμφέροντα, αλλά να υπερασπιστούμε τα αμοιβαία συμφέροντα. Για τις θεωρήσεις, ναι. Όποιο θέλει να έρθει, ένα ελεύθερο κόσμο είμαστε και δεν θέλουμε να μπλοκάρουμε κανέναν. Δεν έχουν κάποιε ανησυχίε. Αλλά υπάρχουν εμπόδια για του Ευρωπαίου που θέλουν να πάνε στην Κίνη, γιατί εκεί δεν πάει οποιοδήποτε. Ούτε και σε οποιοδήποτε μέρο πάει οποιοδήποτε. Καλέ οι σχέσει φιλία, φυσικά όλοι το θέλουμε αυτό. Πρέπει όμω να εμβαθύνουμε. Να ζητήσουμε να διανοίξουν δρόμου ελευθερία και από κοινωνικονική πλευρά και σε ό,τι αφορά τη διέλευση και για του Ευρωπαίου οι Κινέζοι. Αλλιώ ο κινησμό μα πάει πολύ μακριά. Δεν θέλω να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα, αλλά η αμοιβαιότητα δεν πρέπει να μας φοβίζει ως λέξη. Θέλουμε να πάμε στην Κίνα οι Ευρωπαίοι, αλλά να είναι εύκολα τα πράγματα. Να μην μας διαβάζουν τα δικαιώματά μας και τις υποχρεώσεις μας. Και απ' την άλλη να δεχόμαστε με ανοιχτά χέρια και ανοιχτές αγκάλες ε, όλους τους Κινέζους. Δεν θέλω να είμαι κοινικό. Ε, ρεαλιστής θέλω να είμαι. Πρέπει όμως να τα θέσουμε τα πράγματα ω έχουν. Αν θέλουμε να υπάρχουν πραγματικές συνθήκες ε, συμβίωση μεταξύ των δύο πλευρών. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Να σας πω όμως ότι το να μπει κανείς ε, στη... στην Αμερική δεν είναι και τόσο πιο Εύκολο από ότι να πάει στην Κίνα. Πάντως είναι σημαντικό το ερώτημα. Ερωτήσεις άλλες υπάρχουν, τάσεις, αν όχι. Θα παρακαλέσω τον ε, κύριο Πετομάκη. Thank you, Mr. Chair. And... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα. Νομίζω ότι η Κλάουντια Μοντέρο μίλησα για τις θεωρήσεις, μίλησα για τις ε, διατυπώσεις και όταν μιλάμε για βιώσιμο τουρισμό αυτό πρέπει να το δείτε ευρεία τη ενία. Και η περιφερειακή κατανομή. Θέλουμε να είναι στο δυνατόν πιο ευρεία για να έχει αυτό θετικά αποτελέσματα μεγιστοποιημένα και να αποφύγουμε αρνητικές συνέπειες. Και ο κ. Μαντενκάμπ και εσείς μιλήσατε για τις θεωρήσεις διαβατηρίων. Υπάρχει πρόταση από το 2014 για να κώδικα θεωρήσεων. Αλλά υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στα κράτη-μέλη. Τώρα είμαστε στη φάση που προετοιμάζουμε ένα νέο κώδικα. Το ερώτημα είναι τι επίπεδο φιλοδοξία έχουμε. Ελπίζω μέχρι το Μάρτιο να έχουμε τη νέα πρόταση τη Κομισιόν. Και βέβαια συνεχίζονται διμερώς οι συζητήσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Για να είμαι ειλικρινή, δεν νομίζω ότι προβλέπεται ταχεία λύση. Πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά και να δούμε και διμερώς τα πράγματα. Άλλες ερωτήσεις. Σε σχέση και με αυτά που είπε ο Πρόεδρος. Αν αρκεί μια πλήρες χρονιά, είναι καλή αρχή σίγουρα, αλλά μια χρονιά δεν αρκεί. Πρέπει προσπάθειες να είναι συνεχής. Πάντως είναι καλή η βάση αυτή για τη μελλοντική συνεργασία ιδίως οικονομικοί φορείς έχουν αρχίσει σχέσεις και εδώ τίθεται και το θέμα της αμοιβαιότητας. Να είναι πιο εύκολη πρόσβαση στις αγορές ένθεν κακήθεν, τους οικονομικούς φορείς. Αυτό θα ωφελήσει με τον πλέον βιώσιμο τρόπο και τον τουρισμό. Οι εκστρατείες πρόθεσης και προβολής αυτό είναι άλλωστε και ο στόχος αυτής της χρονιάς του ορισμού της Κίνας. Δείχνει και στις χώρες μέλη ποια είναι η προσθέμενη αξία του να γίνονται κάποια πράγματα σε επίπεδο ευρωπαϊκό και όχι εθνικό. Έθεσα κάποιους στόχους, αν τους πετύχουμε αυτό θα πείσει. Και μπορεί αντίστοιχες δράσεις να βρουν μιμητές και στο μέλλον. Η Ινδία την αναφέρατε. Θα ήταν ένα παράδειγμα. Επίσης, οι υποδομές πρέπει να μας απασχολήσουν. Πολύ καλό ερώτημα αυτό για τις υποδομές. Στη χώρα μου Υπάρχει τεράστια ζήτηση για να έρθουν από το Πεκίνο και από όλη την Κίνα να δουν τον Άγιο Βασίλη στη Λαπωνία. όχι ότι και εκεί μπορεί να φιλοξενηθούν πάρα πολλοί Κινέζοι, αλλά προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις υποδομές. Συνολικά είμαστε αισιόδοξοι και νομίζω ότι μπορούμε πια να κάνουμε, αφού σχεδιάσαμε όλες αυτές τις προσπάθειες, να κάνουμε πράξη ε, τους στόχους. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία που έδωσα νομίζω μπορούμε να τα πετύχουμε, αλλά είναι η αρχή μιας μικράς προσπάθειας. Και έχουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα, την αμοιβαιότητα, την πρόσβαση αγορές. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και θα τα λάβουμε και εμείς σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πατομάκη. Λέω πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε όπως σας είπα εδώ ορισμένους ε, συμμετέχοντες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού και Κινέζους συναδέλφους όμως τον Γκόντζιου Φάγκ πρόεδρο το μεγαλύτερο πανεπιστημίο τουρισμού, σχολής τουρισμού και φιλοξενίας και μιλήσαμε και προηγουμένως μαζί για να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τουριστικής Βιομηχανίας και της Κινέζικης Τουριστικής Βιομηχανίας. Στον τομέα των δεξιοτήτων. Και συζητήσαμε και το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις σχολές και τις ακαδημίες ε, κτλ. Αυτό ουσιαστικά το λέω για να καταλάβετε ότι έχουμε και Κινέζους εδώ μέσα στην αίθουσα προσκεκλημένους. Πάμε στο επόμενο σημείο της μεσαίας διάταξης που είναι τα αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 σε σχέση με τον τουρισμό. Τέσσερις ομιλητές. Περιμένουμε τον Γενικό Γραμματέα κύριο Πόλο Λικασβίλη που έρχεται είναι στο δρόμο. Σε κανένα εικοσάλεπτο θα είναι εδώ. Όμω, έχουμε και άλλους ομιλητές που θα προηγηθούν. Πρώτος ο Πιέρ Μπισόφ από τη Eurostat. Ελπίζω να έχετε να μα δώσετε καλά νέα για τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον τουρισμό, τον τουρισμό στην Ένωση το 2017. Έχετε το λόκερ Μπισόφ. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορώ να είμαι σχετικά σύντομος διότι σας μοιράστηκε ένα ενημερωτικό σημείωμα πριν από τη συνεδρίαση, οπότε θα περιοριστώ στα βασικά σημεία αυτού του ενημερωτικού σημειώματος, το οποίο συνετάχθη ε, βάσει του δημοσιευθέντος στον τύπο που έγινε από τη Eurostat για τον τομέα στέγασης του τουρισμού και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία 24 Ιανουαρίου φέτος ημερομηνία δημοσίευσης. Με τα δεδομένα της περσινής χρονιάς. Και να θυμίσω ότι τα δεδομένα αυτά τα συγκεντρώνουν τα κράτη-μέλη ε, βάσει του κανονισμού του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που είχε εγκριθεί από το 2011 τα αποτελέσματα που βλέπουμε για τον τομέα στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017 είναι και πάλι αύξηση. Αύξηση στον αριθμό νυχτών διανυκτερεύσεων που περνάνε οι τουρίστες με 3,2 δις διανυκτερεύσεις 5,2% αύξηση το 17 σε σύγκριση με το 16. Από το 9 λοιπόν παρατηρούμε σταθερή αύξηση στον αριθμό διεκτερεύσεων. Στον τομέα στέγασης δηλαδή των ξενοδοχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των καταλημάτων. Πέρσι είχαμε τέτοια αύξηση στην Λετωνία, τη Σλοβενία και την Κροατία. Στις χώρες αυτές είχαμε αύξηση πάνω από 10% στην εκτερεύσεις. Και σε όλες τις χώρες παρατηρήθηκε αύξηση, εκτός από μία, το Λουξεμβούργο. Η Ισπανία ήταν ο πρώτος προορισμός για τους αλλοδαπούς με την Ιταλία και την Γαλλία μετά. Αυτά για τον αριθμό διενεκτερεύσεων στον τομέα των ε, καταλήμματων. Αυτό έχει συνεισφέρει στον ευρωπαϊκό ισολογισμό, το εμπορικό ισοζύγιο. Και από το 2008 βλέπουμε να υπάρχουν αρκετά περισσότερα ταξίδια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από εκτός από σημεία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό ε, έχει επιβεβαιωθεί ήδη πέρσι από τα τελευταία τρίμηνα του 2017 ε, και μέχρι το τέλος. Και για την απασχόληση στο τομέα του τουρισμού, ενώ ο τουριστικός κλάδος έχει σημαντική θέση στην οικονομία των κρετών μελών, με τις τουριστικές δραστηριότητες να αποτελούν μια μεγάλη ενδυνάμει πηγή απασχόλησης, η απασχόληση στον τομέα των καταλημάτων ε, αναπτύχθηκε και πέρσι με 17% περισσότερη απασχόληση σε σχέση με ένα άλλο ποσοστό του 2008, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στον τομέα του τουρισμού υπάρχει ε, και απασχόληση με ατόμων με χαμηλές δεξιότητες. Για τις πρώτες εκτιμήσεις και τα τουριστικά δεδομένα από πέρσι. Υπάρχει και το ανάλογο website. Θα ενημερώνετε ε, σταδιακά τους ερχόμενους μήνες με αναλύσεις για γεωγραφικά δεδομένα που θα πιο συγκεκριμένα, με αυξητικά και με στοιχεία φθήνοντα και με τα ανάλογες γραφικές παραστάσεις, ώστε να είναι φιλικά προς τον χρήστη. για να δούμε καλύτερα την τουριστική δραστηριότητα της περσινής χρονιάς. Thank you so much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Πετωμάκη τώρα, εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Growth πάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν κοιτάμε τις δραστηριότητες, τις σχετικές με τον τουρισμό, βλέπουμε βέβαια ποια είναι τα αποτελέσματα ή ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον. Η Eurostat δείχνει ξεκάθαρα πως η αντοχή επέδειξε ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση από το 2009 και μετά. Δηλαδή όταν κοιτάει κανείς τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Ο τουρισμός είναι από τους πιο επιτυχείς κλάδους στην Ευρώπη. Με τα τελευταία στοιχεία που βλέπουμε, όντως εντυπωσιαζόμαστε. 500 εκατομμύρια ξένους τουρίστες υποδέχτηκε η Ευρώπη πέρυσι, κάτι που είναι αύξηση 8% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ε, όμως πρέπει να αποκρύψουμε συγχρόνως ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές. Και γι' αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η καινοτομία και οι επενδύσεις στον τουρισμό πρέπει να ενισχυθούν με βιώσιμο τρόπο. Και να μπορούμε επάξια να συμμετέχουμε στο διεθνή ανταγωνισμό. Άρα να στραφούμε προς την Ασία αν θέλουμε να ενισχύσουμε τις τουριστικές ροές και τον ειρηνικό. Να έχουμε νέες αγορές. Σε αυτού του είδους τις πολιτικές χρησιμοποιούμε τη διαφοροποίηση, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα. Αυτά τα τρία είναι πάρα πολύ βασικά και περιγράφουν τι είδους δραστηριότητες θέλουμε, σε τι δραστηριότητες προσβλέπουμε. Και να δούμε Ποιε είναι οι δράσει που έχει στο μυαλό τη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να υπάρξει καλή πλαισίωση των επιχειρήσεων. Έπειτα, ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και περιβάλλον και πώς συγκεκριμένα μπορούμε να έχουμε μια εταιρική σχέση με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και τι οικονομικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην ανάπτυξή τους. Γι' αυτό κοιτάμε και την πλατφόρμα για την ε, έξυπνη ειδίκευση, όπου περιλαμβάνεται και θεματικό τμήμα για τον τουρισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να δούμε πώς θα φτάσουμε στους περιφερειακούς φορείς, στις επιχειρήσεις επιτόπου. Γι' αυτό και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε νέα προγράμματα ιδιωτικών επενδύσεων και χρηματοδότησης. Είναι ζωτική σημασία σε αυτό. Δεύτερον, όπως συμβαίνει και αλλού, έτσι και εδώ, πρέπει το εργατικό δυναμικό να διαθέτει τα προσόντα που χρειάζεται. Και εδώ έχουμε ευρωπαϊκά μέσα το Erasmus Συν, το COSME, με προπολογισμό και μία από τις εμβληματικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν το blueprint για την τομεακή συνεργασία. Στηρίζουμε και το Erasmus Sin, όπως είπαμε, το πρόγραμμα αυτό που βοηθάει αυτή τη συνεργασία. Εκεί ενισχύουμε τα, τη βοήθεια για τα προσόντα που χρειάζεται ο τουρισμός στους υπαλλήλους του. Και προσπαθούμε να βελτιώσουμε και την αντίληψη του, των τουριστικών επαγγελμάτων και να τα παρουσιάσουμε σαν μια ευκαιρία όπως είναι. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον κλάδο να προσελκύσει νέους με προσόντα. Και έτσι όταν πέρυσι είχαμε κάποιες ημερίδες για τις δεξιότητες, συζητήσαμε για τα προσόντα που χρειάζεται ο κλάδος και αυτό συνδέεται και με την ψηφιακή τεχνολογία και τις νέες τεχνολογίες. όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει ανταπόκριση. Τα προσόντα δηλαδή που έχει ο κόσμος στον τουρισμό δεν είναι αρκετά για να ανταποκριθούν σε αυτές τις ψηφιακές προκλήσεις. Έχουμε φροντίσει να ενημερώσουμε και το πόρταλ μας για τον τουρισμό. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες με σεμινάρια και αυτό είναι κάτι πολύ βασικό ως προσέγγιση. Επίσης, η συνεργατική οικονομία και εδώ είναι ένα νέο φαινόμενο, αλλά διευκολύνουμε τις χώρες μέλη για να έχουν ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών προκειμένου να καταλάβουν πώς αυτό το νέο business model μπορεί να τους είναι χρήσιμο και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως και οι παραδοσιακές δραστηριότητες στον τουρισμό. Δεν θέλουμε από την άλλη να κάνουμε τη ζωή των πολιτών μας δύσκολη όταν θέλουν να νοικιάσουν τα διαμερίσματά τους, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται σε σεβασμό απέναντι στην τοπική κοινότητα. Οπότε, συμπληρώνουμε τις προσπάθειες που κάνουν οι χώρες μέλη και οι τρίτες χώρες. Το έτος τουρισμού 2018 και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δίχως άλλο ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς προσπαθούμε να ενισχύσουμε την αμοιβαία αναγνώριση και κατανόηση αλλά και την συνεργασία. Και βέβαια χρειάζεται και διπλωματία. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο, αλλά θέλουμε το διάλογο, να ενισχύσουμε τις επενδύσεις, να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες δηλαδή και για τους Ευρωπαίους και για τους Κινέζους με αμοιβαιότητα και να προωθήσουμε την βιωσιμότητα και την διαφοροποίηση. Ξέρετε τους ευρωπαϊκούς προορισμούς αριστείας, είναι κάτι που οργανώνουμε ήδη από το 2009. Και εκεί αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που γίνονται για την βιωσιμότητα στους λιγότερο γνωστούς προορισμούς, με μοναδικές ευκαιρίες. Ακολουθούμε διάφορα θέματα κάθε χρόνο και φέτος πρόκειται για την πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή θα βραβευτεί η καλύτερη πολιτιστική κληρονομιά που προωθείται μέσω του τουρισμού. Και αυτό γίνεται σε συνεργασία με άλλες γενικές διευθύνσεις. Πιστεύουμε ότι η εταιρική σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα για την προώθηση του τουρισμού και διακρατικά αλλά και διαπεριφοριακά είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Κάτι άλλο για το 2018 είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Εφιούς Τουρισμού. Το γνωρίζει και ο πρόεδρος πολύ καλά. Με τη δράση αυτή θα δώσουμε βραβεία στις πόλεις που κάνουν ιδιαίτερες προσπάθειες για να προσφέρουν τις καλύτερες εμπειρίες στους επισκέπτες τους, μέσω ψηφιακών εργαλείων επίσης. Και θα έχουμε και ένα πλαίσιο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων προορισμών. Και τέλη Μαρτίου θα αρχίσει και στο σελίδα μας με πρωτοβουλία που θα ζητήσει από τις ε, ευρωπαϊκές πόλεις να είναι υποψήφιες για το βραβείο εφίους τουρισμού για το 2019. Κάποια άλλα σημεία τώρα. Για το 2018 είναι η χρονιά πολιτιστικής κληρονομιάς. Μεγάλη ευκαιρία για τον ευρωπαϊκό ε, τουρισμό και πολιτισμό. Θα έχουμε διάφορες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις. Στηρίζουμε προσπάθειες για αριστεία στις διάφορες ευρωπαϊκές περιοχές με βιώσιμο τρόπο και καινοτομία πάντα με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το οποίο συνεργαζόμαστε, όπως επίσης και με την UNESCO, για να προωθήσουμε τα προγράμματα εκείνα τα οποία προάγουν την πολιτιστική μας κληρονομιά στα πλαίσια του τουρισμού. Με κονδύλια από το κόσμο, επίσης για το θεματικό τουρισμό. Και τέλος, ασφάλεια, τουρισμός και ασφάλεια. Όλοι γνωρίζετε ότι πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σύστημα αίτιας με στόχο να ενισχύσει την ασφάλεια αλλά και να διευκολύνει τα ταξίδια χωρίς θεωρήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι βλέπουμε πολλές ευκαιρίες να παρουσιάζονται στον κλάδο του τουρισμού. Τα στοιχεία τα νούμερα που μα ήρθαν από τον Eurostat είναι μια σαφής ένδειξη για το ότι δεν έχουμε φτάσει στα όρια της ανάπτυξης. Μπορούμε δηλαδή να εκμεταλλευτούμε περισσότερες ευκαιρίες Εμείς προσφέρουμε το σωστό πλαίσιο και εκεί μέσα μπορούν να αναπτυχθούν πολλές δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τον τουρισμό μας. χρησιμοποιώντας πολλά μέσα και υποφελούμενοι από καινοτομίες και βιωσιμότητα στην οικονομία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η επόμενη παρουσίαση από τον Εντουάρντο Σανταντέρ. Έχετε και εσείς μερικές διαφάνειες βλέπουμε. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου, κύριε Πετομάκη, συνάδελφοι από τη ΓΑΜΑ τη Μάνα του Ευχαριστώ που με προσκαλέσετε και εμένα σήμερα. Θα ήθελα και εγώ να σας δώσω κάποιες πληροφορίες μετά από τα στοιχεία που έδωσε ο συνάλφος της Eurostat και θα σας ε, δώσω και μια ερμηνεία για το τι συνέβη το 2017. Ξεκινώ με καλά νέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο ε, ανθούσες περιφέρειες και ελκυστικούς προορισμούς. Το 2017 ήταν ε, ε, μία καλή χρονιά. Η αύξηση που παρατηρήθηκε κάλυπτε περισσότερους προορισμούς. Πάνω από 5% έχει μέρη αγοράς η Ευρώπη και πάνω από 650 εκατομμύρια τουρίστες έφτασαν το 2017. Αυτός ο αριθμός μεταφράζεται σε ένα 8% αύξηση σε σχέση με το 2016. Για όδο συνεχόμενο έτος κατακυρώθηκε ότι η Ευρώπη είναι βασικός τουριστικός προϋπολογισμός και και στις ε, μεγάλες αποστάσεις και στις ε, ενδοκινοτικές τουριστικές αγορές. Το 5% του τουρισμού είναι ακόμη εγχώριος, ε, ευρωπαϊκός δηλαδή. Επίσης, υπήρξαν κάποια προβλήματα ασφάλειας και αυτό είχαμε και ιδίως στη, σε Βέλγιο, Γαλλία και Ισπανία στροφή στον εσωτερικό τουρισμό. Θα τα πούμε και για τις υπεράκτης περιοχές. Είχαμε αύξηση ουσιαστικά σε όλους ε, τους ε, προορισμούς που παρατηρήσαμε. Πάνω από η μισή από αυτούς ε, έχουν αύξηση διψήφια, πάνω από το 10%. Δυτική Ευρώπη. Μετά από χρόνια ύφεση λόγω των πολιτικών αναταραχών και ανασφάλειας και με τον Brexit ε, άλλαξα η κατάσταση λοιπόν. Είναι μεγάλη αύξηση της Ανατολικής Ευρώπης στα συνολικά νούμερα. Όμως ο βασικός ε, νικητής πια πέρσι ήταν ε, η Νότια Μεσόγειος. Μάλτα, Σλοβενία, Κύπρος και Ισπανία σημείωσαν ρεκόρ. Μιλάμε επίση για το έτος τουρισμού με την ε, Κίνα και θέλω εδώ σε αυτήν την διαφάνεια να σας ε, πω πόσο σημαντικές είναι αυτές οι μακρέ μακρές αποστάσεις. Ε, το 2017 βελτιώθηκαν τα πράγματα σε με το 2016. Κίνα, Ιαπωνία, ανατολική Ασία, Βόρεια Αμερική που είχαν πληγεί σημαντικά σημειώνουν μια ανάκαμψη το 2017. οικονομική ανάκαμψη θα συνεχιστεί το 2018 στις περισσότερες από αυτές τις βασικές αγορές. Συνολικά οι ευρωπαϊκές αφήξεις έχουν φτάσει σε νέα ύψη το 2017. Από Ρωσία, τουριστικές ροές συνεχίζουν να ανακάμπτουν μετά από μια σειρά ετών που δεν είχαμε τέτοια θετικά στοιχεία. Η Ρωσία ξανάρχεται. Οι Ρώσοι ξανάρχονται, αγαπητοί συνάδελφοι. 15 εκατομμύρια αφήξεώσαν το 2017, 7% αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι Αμερικανοί ωφελούνται λόγω του ισχυρού νομίσματος και ανταγωνιστικά έχουν το πλεονέκτημα. Το 2017 είχαμε αύξηση 12%. Ξεκολουθούν να προτιμούν την Ευρώπη σε σχέση με άλλους προορισμούς. Οι Αμερικανοί, είπα, είναι και ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος ε, ε, χώρος από τον οποίο έρχονται οι τουρίστες ε, στην Ευρώπη. Βελτιώθηκαν επίσης οι αεροπορικές συνδέσεις με την Κίνα. Ε, το θέμα της συνδεσιμότητας είναι ένα θέμα, το ανέφεραν. Άρα με την Κίνα έχουμε εδώ βελτίωση. Και η μεσαία τάξη αυξάνεται, άρα θα αυξηθούν ε, και οι τουρίστες από αυτή την περιοχή. Το 2017 είχαμε 12 εκατομμύρια Κινέζους επισκέπτες. 16% αύξηση σε σχέση με το 2016. Υπάρχει δυναμικό, ναι υπάρχει. Είναι βιώσιμο αυτό το δυναμικό. Αυτό είναι και το ερώτημα. Νομίζω ότι αυτό το τουριστικό έτος μπορεί να μας δώσει λύσεις. Ινδία. Μικρή αγορά, αλλά είναι πολλά υποσχόμενη. Το 17,26 εκατομμύρια αφήξεις καταγράψαμε από την Ινδία που θα γίνει όλο και περισσότερο μια σημαντική αγορά. Ερωτηματικό εδώ και για την προώθηση, προβολή και τις επενδύσεις. Συνολικά το θετικό αποτέλεσμα το περιμένουμε και για το 2018, αύξηση δηλαδή. Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από τους οικονομικούς φορείς, και νομίζω ότι και το κόστος ακόμη και αν αυξηθεί δεν θα αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα. θετικές οι προοπτικές ε, ε, μετάσεις ε, για αύξηση της ανάπτυξης κατά 4%. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που συνηγορούν στο να είμαστε βασικός τουριστικός προορισμός. Η ισχυρή συνεργασία μεταξύ των προορισμών και των διαφόρων μπλεκομένων διαφοροποίηση του μείγματο επισκεπτών και σωστή στοχοθέτηση επισκεπτών εκτός των δεσποζωσών ε, αγορών. Δηλαδή και αναδυόμενες και σταθερές αγορές παραδοσιακές. Πρέπει επίσης να αυξηθεί η ανθεκτικότητα και η τουριστική ανάπτυξη. Για να γίνει αυτό χρειάζεται συνεργασία μεταξύ τουριστικών προορισμών και τουριστικών φορέων. Για να υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση αν θέλουμε να αναπτυχθεί μακροχρόνια και βιώσιμα ο τουρισμός. Με την ανάκαμψη ανοίγει ο δρόμος ε, ώστε οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές να στραφούν στην ανάπτυξη του τουρισμού, της βιώσιμης ανάπτυξης ε, να είναι καταλήτης ο τουρισμός και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τέλος, συνεργασία είναι σημείο κλειδί. Είχαμε μία ε, πρωτοβουλία με το μανιφέστο για τον τουρισμό για να δείξουμε ότι ο τουρισμός ε, όχι απλά τώρα έχει σημασία, αλλά θα συνεχίσει να έχει σημασία και στο μέλλον. Νομίζω ότι με αυτά σας έδωσα κάποιες ιδέες για το πού πηγαίνουμε και για το από πού ερχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, Εντουάρντο. Και πρέπει να πούμε ότι η παρουσίαση της ε, Επιτροπής, της Eurostat, είναι κάτι για το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε. Μπορεί να έχετε ερωτήσει. Έχει ζητήσει το λόγο ο συνάδελφος, ο κύριος Δεγκράντες Πασκουάλ επίσης, ε, είναι διάφοροι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο και εντωμεταξύ ίσως να έρθει και ο Γενικός Γραμματέας. Ο κύριος Βαντερκάμπ. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στη Eurostat και ευχαριστώ. Τους πίνακες που μας έστειλε και μας παρουσίασε ε, βρίσκω ότι είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικοί. Η ερώτησή μου είναι, κύριε Σανταντέρ, αν και απάντησε σε ένα βαθμό, ο βελγικός και ο γαλλικός τουρισμός έχει επιστρέψει στα παλιά επίπεδα, αυτό είπατε, πριν τις επιθέσεις. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, ο τουρισμός δίνει πολλές ευκαιρίες σε ανθρώπους που δεν είναι ιδιαίτερα μορφωμένοι, είναι σε, μισέ, σε μεσαία επίπεδα μόρφωσης. Σωστή παρατήρηση. Τι δηλαδή ευκαιρίες για δουλειά προσφέρει ο τουρισμός σε προσωπικό τέτοιας μεσαίας κατάρτισης. Πολύτιμο αυτό. Και τώρα για τον κύριο Σανταντέρ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει αρκετά από πλευράς πολιτικής τουρισμού, κατά τη γνώμη σας. Και θέλουμε βέβαια να είσαστε ειλικρινείς στην απάντησή σας, έτσι. Πρώτα να ε, κάνει την ερώτησή του και ο κύριος ε, Πασκουάλ, την Γκράντες Πασκουάλ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο πράγματα. Πρώτον, όπως και ο συντονιστής μου, Βαντερκάμπ, και εγώ κρατάω κάποια πράγματα που είπε η Eurostat για τη δημιουργία απασχόλησης για ανθρώπους ε, όχι ιδιαίτερα υψηλής κατάρτισης. Ο τουρισμός δηλαδή δημιουργεί θέσεις απασχόλησης που πολλές φορές δεν είναι πολύ μόνιμες σε εστιατόρια, καφετέριες. Στην Ισπανία είναι κάτι που το γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί έχουμε τεράστιο τουρισμό, παγκόσμια ρεκόρ, αλλά που βέβαια κυμαίνεται δεν είναι πάντα μόνιμες οι θέσεις απασχόλησης στον τουρισμό. Οπότε η ερώτηση προς τον κύριο Σαταντέρ για παράδειγμα είναι αυτό που ρωτούσε και ο κύριος Βαντερκάμπ. Δηλαδή σε ένα χώρο όπως είναι ο τουρισμός οι αρχές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μέσα ώστε να μειώσουν την εποχικότητα. Οπότε αυτή η αστάθεια που υπάρχει στην απασχόληση στον τουρισμό να μειωθεί. Πρέπει να βρούμε πολλούς τρόπους, πολλά εργαλεία ώστε η απασχόληση αυτή του τουρισμού να γίνει πιο μόνιμη και να μπορούν οι διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις να ζουν ολόκληρο το χρόνο από τον τουρισμό. Έπειτα και τη συνεργατική οικονομία. Ναι. Υπάρχουν πόλεις όπως είναι η Βαρκελόνη που υποδέχεται πάρα πολλούς τουρίστες και έχουμε φτάσει σε αυτό που ονομάζουμε τουρισμοφοβία. Και γιατί. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί τα διαμερίσματά του και παράνομα τα ποινικιάζει κάνοντας αθέμητο ανταγωνισμό στα ξενοδοχεία, όπως καταλαβαίνετε, για να κερδίζουν ε, χρήματα χωρίς να τα δηλώνουν. Εντάξει, οπότε τι είστε το θέμα, ποιος πληρώνει φόρους, ποιος δεν πληρώνει. Και γι' αυτό όσοι πληρώνουν φόρους και νόμιμα νοικιάζουν διαμαρτύρονται για τις άλλες μορφές ε, ενοικίασης που δεν είναι επίσημες. να υπάρχει και κοινωνικός τουρισμός, αλλά να μην υπάρχει αθέμετος ανταγωνισμός όπως υπάρχει σήμερα από αθέμετες τέτοιες πρακτικές. Εγώ δεν θέλω εδώ να αναφερθώ σε καμία επιχείρηση, αλλά είναι κάτι που πρέπει να αναλύσουμε περισσότερο ό,τι έχει να κάνει με τη συνεργατική οικονομία. Ευχαριστούμε κυρία Μοντέρο πολύ γρήγορα, γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε και χρόνο. Απλώς αυτό το γύρο των ερωτήσεων προς τον Εντοάρντο, να προσθέσω κι εγώ. Τι είδου δράσεις συγκεκριμένα προβλέπονται για φέτος. Και πώς προβλέπετε να μειωθεί, να ανακατανεμηθεί το σκέλος της προώθησης πώς θα προβάλλουμε τους πλέον γνωστούς προορισμούς και τι έχετε κατά νου για να γίνει αυτό. Και ως προς την πλατφόρμα των επενδύσεων για την προώθηση των τουριστικών σχέσεων Ευρώπης-Κίνας, μπορείτε να μας πείτε πώς έχει το state of play αυτής της πλατφόρμας. Ευχαριστώ. Ε, Jill Evans, Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, όπως και να δούμε τα στατιστικά στοιχεία και ε, με συγκεκριμένο τρόπο να λάβουμε γνώση των ε, μετακινήσεων και το τι αντίκτυπο έχουν στην οικονομία της θέσης απασχόλησης και το τι μελλοντικές εξελίξεις προβλέπονται. Εγώ εκπροσωπώ την Ουαλία, όπου ο τουρισμό ε, αναπτύσσεται γοργά και έχουμε υποφεληθεί ιδιαίτερω ε, στην οικονομία μα. Ε, Όμω, ω προ τα, τα στατιστικά, συχνά συζητούμε σε αυτό το φόρουμ ε, την προσβασιμότητα και με ενδιαφέρει να μας πείτε αν υπάρχουν δεδομένα για την προσβασιμότητα των ανθρώπων που έχουν μειωμένη κινητική, κινητικότητα. Όχι μόνο στα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία, αλλά και σε μουσεία, και σε άλλα αξιοθέατα. Δηλαδή να κοιτάξουμε η ανάπτυξη του τουρισμού να εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων. Ευχαριστούμε. Εγώ θα θέσω την τελευταία ερώτηση μόνος μου προς τον Εντουάρντο Σαντάντερ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η στον ήτηση σε άλλους ε, φορείς. Κοιτάζει κανείς τις συνέπειες ή τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει το Brexit. Βλέπουμε τους αριθμούς του 2017 αλλά και αυτό να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε δεν μπορεί να γίνει σε 2-3 χρόνια. Η Επιτροπή Μεταφορών έχει ε, ασχοληθεί με τις ε, συνέπειες του Brexit στον τομέα των μεταφορών. Στον τομέα του τουρισμού τι προβλέπετε, υπάρχει κάποια γνώση για το τι μπορεί να γίνει. Έχετε κάποια σχετική πληροφορία. Θα μας απαντήσω, ο κύριος Μπίσοφ από την Eurostat. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για την παρουσίαση που μας αφήσατε να κάνουμε από την πλευρά της Eurostat, Βέλγιο και Γαλλία. Ε, εκεί παρατηρήθηκε ανάκαμψη του τομέα του τουρισμού μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Η απάντησή μου λοιπόν θα ήταν καταφατική, αλλά συγχωρέστε με δεν έχω μαζί μου τους αριθμούς. Ε, σας προτείνω να σας τα αποστείλω. Θα σας στείλω ακριβέστερους αριθμούς για το πόσο μεγάλη ήταν η ανάκαμψη. Στην ερώτηση του συναδέλφου σας για τα στατιστικά, και την προσβασιμότητα. Φοβούμε ότι πολύ λίγα γνωρίζουμε. Και πάλι δεν έχω ακριβείς αριθμούς αλλά θα μπορούσαμε να τα διασταυρώσουμε από διαφορετικές πηγές δεδομένων, ξέρω εγώ, ε, το εργατικό δυναμικό, τις συνθήκες διαβίωσης και το εισόδημα και μπορεί να προκύψουν ενδιαφέροντα στοιχεία ακόμη και, αν, και πάλι δεν πιστεύω ότι θα έχουμε για πάρα πολλά αλλά μπορούμε να τα στείλουμε στη γραμματεία της Επιτροπής ό,τι διαθέτουμε στις βάσεις δεδομένων μας και μετά έγινε μια παρατήρηση για τις χαμηλές δεξιότητες και την παραγωγικότητα στον τουριστικό κλάδο. Ίσως δεν είναι δουλειά της στατιστικής υπηρεσίας να απαντήσει σε αυτό. Νομίζω αυτές ήταν οι ερωτήσεις που απευθύνονται σε μένα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σας ευχαριστούμε. Από την Επιτροπή κύριος Πεταλμάκη. Ναι, ναι, δεν θα απαντήσω εγώ για τον κύριο Σαββαντέρ. Θα του αφήσω να απαντήσει μόνο του τι ερωτήσει του. Θα μα πει αν κάνουμε αρκετά ή όχι άλλωστε. Ε, σω πιο συγκεκριμένα για τι δεξιότητε. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που απασχολεί όχι μόνο προς τον τουριστικό κλάδο, αλλά συνολικά. Βλέπουμε την τεχνητή ευφυία, τη ρομποτική, πολλές παραδοσιακές θέσεις εργασίας που χάνονται. Ή υποκαθίστανται από κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με αυτές τις δουλειές που απομένουν. Υπάρχει ανάγκη για διαφορετικό είδος υπηρεσιών και άλλη μορφή εργασίας, θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει να δούμε τι τομεακέ δεξιότητε στα πλαίσια τη ατζέντα μα για τα επόμενα χρόνια και προσπαθούμε να έχουμε μια ευρεία διαβούλευση με του ενδιαφερομένου για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε τομεακή βάση. Ξέρετε ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά τη αγορά εργασία. Πάντω υπάρχουν συγκεκριμένε ανησυχίε που είναι δικαιολογημένε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι ιδιαιτερότητε που αναφέρατε και εσεί. την οποχικότητα, το χρόνο, την εργασία μερικού χρόνου. που, στοιχεία που μπορεί να εμποδίζουν την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, ε, ξέρω εγώ, τα, τις συμβάσεις σύντομες προσπαθούμε αυτά να τα διασταυρώσουμε με το τι δουλειά θα μπορούσε να γίνει για να αναπτυχθεί το σύνολο δεξιοτήτων που θα ήταν χρήσιμα κάτι που να είναι πιο ε, κατάλληλο, πιο ευστοχό για τους νέους και ταλαντούχους, για τον τουριστικό κλάδο, να το προσελκύσουμε εκεί. Συνολικά, αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σε όλο το εύρος των οικονομικών μας ε, δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης. Όταν μιλάτε για συνεργατική, για συμμετοχική, ε, για οικονομία, Πρέπει να σκεφτούμε πώς αλλάζουν τα κλασικά επιχειρηματικά μοντέλα και αν μπορούμε ως πολιτικοί ηθήνοντες, αυτοί που σχεδιάζουν την πολιτική, να εξασφαλίσουμε ισότιμους κανόνες παιχνιδιών μεταξύ των διαφορών φορέων στον, ε, στην αγορά εργασία. Για την προβολή των λιγότερων εκπροσωπούμενων περιοχών, εδώ νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα πρόθεσης και ίσως τώρα, Εάν κοιτάξετε τι κάνουμε στο έτος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας 2018, ε, είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι ο καθένας μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα ευρωπαϊκής σε εργαλεία και πλατφόρμες για να προωθηθεί εθνικός, περιφερειακός, τοπικός τουρισμός στο ανάλογο επίπεδο. Όλα αυτά νομίζω ότι ήδη εξελίσσονται για το Brexit Έχουμε εργαστεί σκληρά για να μπορέσει η ομάδα δράσης να έχει στα χέρια της τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάλυση και τη μελέτη του τι αντίκτυπο θα έχει το Brexit. Στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για το πού στοχεύουμε και το τι είδους μελλοντικέ σχέσεις διαβλέπουμε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Να γιατί ε, πρέπει να προχωρήσει η χαρτογράφηση, να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε έναν κατάλογο στοιχείων που θα χάσουμε. Πρέπει να δούμε τις μελλοντικέ σχέσεις βάσει των στόχων που θέλουμε να υπάρχουν μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είμαι και σε θέση να πω περισσότερα. Eduardo Άνετο ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαντενκάμπ. Είναι επίμαχο το θέμα. Απάντοντας απόλυτα ειλικρινά, είναι ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά από την Κομισιόν με βάση το 176β το άρθρο συνθήκησε κάνουν ακριβώς ό,τι πρέπει με πολύ λίγα άτομα και πολύ ε, λίγο προσωπικό. Ο οργανισμός τουρισμού. Τώρα, τι κάνει η Κομισιόν ε, συνολικά, λίγα. 10% το άεπνο τουρισμός. 25 εκατομμύρια θέσει εργασίας δημιουργεί. Δεν το λαμβάνει υπόψη η Κομισιόν όμως σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω και αυτό συζητείται τώρα, ότι θα γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις στην επόμενη νομοθετική περίοδο. Ελπίζουμε, εγώ δεν προσωπώ μόνο το ΕΤΙΣ εδώ, αλλά και τις ενώσεις στις Βρυξέλλες και όλους τους εμπλεκομένους. Θεωρώ ότι οι Βρυξέλλες πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, ως βιομηχανία τον τουρισμό, άρα πρέπει να έχει σημασία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εδώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πέραν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν με επιτρέπετε να απαντήσω στα ισπανικά στον κύριο Ντεγκράντες για την εποχικότητα. Πράγματι. Έχει μεγάλη σημασία για το έτος τουρισμού μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, διότι ο Κινέζος ε, ταξιδιώτης δεν ταξιδεύει όταν ε, υπάρχουν προβλήματα χωρητικότητας, δυναμικότητας, ε, αλλά όταν ε, έχουν την κινέζικη πρωτοχρονιά οι Κινέζοι που τέλειωσε το Φεβρουάριο προηγούμενη και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το φθινόπωρο τέλος πάντων. Αυτό είναι μια μεγάλη ε, ευκαιρία εμάς ε, στην Ισπανία από το Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο λειτουργεί ε, η σεζόν, έχουμε καλοκαίρι. Οπότε αυτό μπορεί να είναι πολύ θετικό για να προσελκύσουμε ταξίδες από τρίτες ε, χώρες, από την Κίνα και άλλες χώρες της Ασίας, από την Ινδία και αυτοί αυτό θέλουν να ταξιδέψουν και σε χώρες που δεν θα βλέπουν μόνο Κινέζους, παραδείγματος χάρη, εκεί που θα πάνε. Υπάρχει και ένα πρόβλημα οργάνωσης σε επίπεδο stakeholders. Θα μπορούσαμε ευρωπαϊκά να δούμε ε, τις σχολικές διακοπές, για παράδειγμα, ανάλογα με τη χώρα. Να τις οργανώσουμε διαφορετικά. για την τουριστική σεζόν, ιδίως για τα Χριστούγεννα και για το καλοκαίρι, ώστε να υπάρξει παράταση της σεζόν δύο-τρεις εβδομάδες. Και αυτό μπορεί να αυξήσει τις συμβάσεις εργασίας και, τον τουριστικό, και τις τουριστικές ροές. Για τη οικονομία εμείς δεν έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρισμού ε, λόγους για να είμαστε περικατά. Η συνεργατική οικονομία για κάποιες χώρες της Ένωσης όπως η Μάλτα, η Ιρλανδία είναι λύση στο πρόβλημα χωρητικότητας, δυναμικότητας, γιατί ενώ υποδέχεται πολλού τουρίστες δεν έχει επαρκείς κλίνες. Απλά θέλουμε να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή. Και τώρα ξαναμιλάω αγγλικά, γιατί θέλω να μιλήσω στην κυρία Μοντέρο. Σε ό,τι αφορά προβολή λιγότερο γνωστών ε, προορισμών σε περιοχές. Hidden Track Destination αυτό το έτος το τουριστικό Κίνα σε Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους προορισμούς θέλει να καλύψει. Όχι Παρίσι, Βαρκελόνη, Ρώμη, Βενετία έχουν διάσημους προορισμούς, αλλά τις ροές αυτές των Κινέζων θέλουμε να τις ε, διοχετεύσουμε σε προορισμούς με τους οποίους δεν είναι εξοικειωμένοι ακόμα. Δεν θέλουμε μόνο να του προσελκύσουμε και να του εξηγήσουμε τι πρέπει να προσφέρουν στα εδάφια αυτά, δηλαδή που του προσελκύσουν, αλλά θα πρέπει να του εκπαιδεύσουν για να ε, φροντίσουν για τους Κινέζους αυτούς ε, επισκέπτες με το σωστό τρόπο, γιατί δεν υπάρχει ακόμη αντιστοιχεία. Και η προσβασιμότητα είναι ένα θέμα, γιατί πρέπει να φτάσουν σε αυτούς τους λιγότερο γνωστούς ε, προορισμούς οι Κινέζοι, αλλά χρειάζεται και κάποια εταιρεία να τους μεταφέρει. Στη χώρα μου υπάρχουν ε, πολλά αεροδρόμια που δεν χρησιμοποιούνται όμω με το σωστό ή επαρκώ. με το σωστό τρόπο επαρκώ. Άρα θα πρέπει να διοχετεύσουμε τι ωραίε αυτέ. όλα τα αεροπλάνα που έρχονται από την Ασία σε δεύτερους προορισμούς, όχι τους τόσο γνωστούς. Η έρευνα αγορά λέει τώρα ότι οι Κινέζοι δεν ενδιαφέρονται πλέον να κάνουν ουρά μπροστά από τον πύργο του Άιφελ ή να βλέπουν ε, άλλους Κινέζους ε, ε στη μίζωνες σε αυτούς τουριστικούς ε, αλλά θέλουν να κάνουν ένα άλλο είδος ε, διακοπών. Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα, είναι μείζον ζήτημα. Εμείς συνεργαζόμαστε και με το Αμαντέους. Δημιουργήθηκε, μάλλον χθες είχαν μια έκθεση, πέρυσι μια έκθεση για την προσβασιμότητα δεν είναι όμως πρόβλημα, αλλά πρόκληση, ευκαιρία. Ένα δις δεν έχουν προσβασιμότητα, καμία. Και δεν μιλάμε για αναπηρία όταν μιλάμε για προσβασιμότητα. Μιλάμε για οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένους, δεγενειακή, δεγενειακά ταξίδια. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη. Και αν συγκρίνουμε άλλε αγορέ, όπως τη ΣΥΠΑ, που εδώ και χρόνια ασχολούνται με τον προεδάσιμο τουρισμό. Όχι ηθικό, αλλά επιχειρηματικό. Γιατί είναι μια τεράστια αγορά αυτή. Τέλος για το Brexit, το μόνο που μπορούμε να πούμε για το Brexit μέχρι στιγμή είναι ότι επηρεάζει την αντίληψη σε τρίτες αγορές για την Ευρώπη όσο πιο πολύ δυσκολέψουμε τη, τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, τα διπυρωτικά, τόσο πιο δύσκολα θα λαμβάνονται και αποφάσεις για, και θα επιλέγονται λιγότερο οι ευρωπαϊκοί προορισμοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει ε, φοβερά επαγγελματικό επίπεδο. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Ο Εντουάρδο ήξερε ακριβώς πόσο χρόνο μπορούσε να μιλήσει, ε, πόσο χρόνο να απαντήσει, ώστε να πετύχει ακριβώς την κατάλληλη στιγμή να σταματήσει όταν έφτασε ο κύριος ομιλητής μας που είναι γενικός γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τον Τουρισμό. Καλώς ήρθατε λοιπόν κύριε Πολιολικασβίλη στην ε, Task Force της Επιτροπής Τουρισμού. Τι θέλετε να ακούσετε. Αγγλικά είναι το νούμερο 2. Λοιπόν, σας καλωσορίζω, έλεγα, Γενική Γραμματέα, του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τον Τουρισμό. Αν υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια τουρισμού στον κόσμο, σίγουρα αυτός είναι ο πατέρας της. είναι ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του ΟΙΕ λοιπόν για τον τουρισμό και ασχολείται με όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Συμφωνήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα και με τον κύριο Σόμοντι ότι θα έπρεπε οι δεσμοί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον οργανισμό αυτό του Ηνωμένων Εθνών να γίνουν πιο στενοί. Και ο νέος Γενικός Γραμματέας τώρα, ο οποίος ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου, εξελέγει πέρυσι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχή που βρήκε το χρόνο, παρά το ότι είναι πολύ άσχολος, να έρθει σε αυτήν την task force της Επιτροπής Μεταφορών. Και αύριο σίγουρα θα είσαστε όλοι παρόντας στην ειδική εκδήλωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθημερινά υπογράφει διάφορες συμφωνίες με οργανισμούς. Τις υπογράφει ο πρόεδρος Ταγιάννη. Αύριο ο πρόεδρος Ταγιάννη και ο γενικός γραμματέας Πολυολικασβήλη θα υπογράψουν ένα μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κάτι πολύ σημαντικό για τον τουρισμό. Ευχαριστούμε λοιπόν και χωρίς άλλη καθυστέρηση σας δίνω και το λόγο. Πέντε ώρα θα πρέπει να ολοκληρώσουμε ή αλλιώς θα συνεχίσουμε χωρίς διερμηνία μετά τις πέντε. Βέβαια και αύριο θα είσαστε εδώ, οπότε θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να σας δούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή. Έφτασα όμως επιτέλους. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία αυτή ευκαιρία που μου δίνετε και χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Όντως, όπως είπατε, είναι ο δεύτερος μήνας που έχω αναλάβει τα καθήκοντά μου από 1η Ιανουαρίου. Και ήθελα να έρθω στις Βρυξέλλες ήδη τους πρώτους μήνες της θητείας μου. έχουμε και στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, σχετικές εκδηλώσεις. Λοιπόν, ο τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός κλάδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη, που παραμένει ο κατεξοχήν προορισμός στον κόσμο, τουριστικός προορισμός. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το αποτέλεσμα που φάνηκε δηλαδή το 2017 ήταν ο κατεξοχήν τουριστικός προορισμός. Τώρα, αγαπητά μέλη της Task Force αυτής, ο κύριος Σταγιάννη το είπε ότι η Ευρώπη είναι πολύ ανταγωνιστική και σε αυτό το τομέα και είναι καλό να βάλουμε από κοινού τις δυνάμεις μας. Και εγώ ήρθα εδώ σήμερα γιατί ξέρω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για ένα κοινό όραμα. Έχει επιτευχθεί πρόοδος, αλλά μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερο για να ενισχύσουμε τον τουρισμό και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Φέτος είναι η χρονιά τουρισμού, είπαμε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και είναι αφιερωμένη στη πολιτιστική μας κληρονομιά. Μετά την υπογραφή του μνημονέου της τελετής θα συναντηθούμε και πάλι με τους Κινέζους εταίρους. Η Κίνα είναι η πιο σημαντική αγορά. Θα παρουσιάσω και εγώ το όραμά μου και τα σχέδιά μου για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Θα επικεντρωθούμε περισσότερο στη βιωσιμότητα των δυνάμεων, που είναι προτεραιότητα για τον οργανισμό τουρισμού του ΟΗΕ. Τεχνολογία, Έχουμε πολλά σχέδια και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί. Η συμμετοχή σας, οι επαφή σας, η στήριξή σας είναι πολύ σημαντικά πράγματα για μας. Τουρισμός και ασφάλεια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα πάνω στο οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ μαζί. Έχουμε διάφορα προγράμματα μπροστά μας. Αρχίσαμε ήδη με τη στήριξη της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Η εκπαίδευση είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του κλάδου. Και αυτό φάνηκε σε εκδήλωση που έγινε για τον τουρισμό με 45 υπουργούς και όλοι είπαν πόσο σημαντική είναι η κατάρτιση σε αυτό το κλάδο. Θα ανοίξουμε λοιπόν διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα. Και μάλιστα μια πρόταση έγινε από την Ουγγαρία όταν συναντηθήκαμε με τον Ούγγρο Υπουργό και θα ανοίξουμε ένα τέτοιο κέντρο εκεί. Πρέπει να ενισχύσουμε επίσης τους δεσμούς του οργανισμού του ΟΗΕ με τις διάφορες χώρες και να ενισχύσουμε και τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, startups και άλλους που προσφέρουν τεχνολογία. Για τα startups θα στηρίξουμε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παντού στον κόσμο και αναχώρα θα αναπτύξουμε προγράμματα για να χρηματοδοτήσουμε τέτοια προγράμματα υπέρ των startups και των νέων τεχνολογιών. Το ωφέλη είναι για όλους μας. Η προτεραιότητα αυτή σημαίνει ότι πρέπει να φροντίσουμε να βρεθεί ακόμα περισσότερο ο τουρισμός θέλουμε να στηρίξουμε την περιφερειακή ολοκλήρωση για νέα προϊόντα και τη συνδεσιμότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι πιο ανταγωνιστική στηρίζοντας την περιφερειακή ολοκλήρωση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις κατάλληλες μεταφορές και άλλα δίκτυα. Χρειαζόμαστε καλές ε, ταξιδιωτικές εμπειρίες τουρίστες εκτός Ευρώπης όταν αποφασίσουν σε ποια ήπειρο θα πάνε, το κάνουν πολύ περισσότερο ανά ήπειρο παρά ανά χώρα. Και γι' αυτό και το θέμα των μεταφορών συνολικά πρέπει να μας απασχολήσει. Κάτι άλλο είναι τα νέα business models. Η νέα πλατφόρμα υπηρεσιών τουρισμού η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί στις αλλαγές με τις κατάλληλες ρυθμίσεις και υπεύθυνα. Έτσι κι δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους, από την άλλη όμως πρέπει να υπάρχει μια ισοτιμία στην αντιμετώπιση. Μπορούμε έτσι να ενισχύσουμε την ποιότητα, την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισμών. Το τρίτο μου θέμα είναι το εξή. Πρέπει να διαχειριστούμε τον μεγάλο αριθμό τουριστών που συγχρόνως φτάνουν σε ένα προορισμό. Το είδαμε αυτό τα τελευταία δύο χρόνια. Φροντίσαμε για την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα αλλά είδαμε ότι μερικές ευρωπαϊκές περιοχές υποφέρουν από αυτό τον υπερβολικό τουρισμό ή μάλλον την υπερβολική συγκέντρωση τουριστών ε, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Πρέπει όμως αυτά να τα αντιμετωπίσουμε κατά περίπτωση και να υπάρξει μια συνειδητοποίηση των ε, ωφελών από τον τουρισμό και ίσως να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα κάνει συστάσεις για το πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Δεν θέλω να μιλήσω για πρόβλημα. Θέλουμε να στηρίξουμε τις πόλεις για να διαχειριστούν τέτοιες ροές τουριστών. Και πρέπει να διαχειριστούμε και τις επιπτώσεις των τουριστικών ροών να προωθήσουμε τουριστικές εμπειρίες από τις οποίες μπορούν να υποφεληθούν άμεσα κοινότητες. Έχουμε ευκαιρίες για ενίσχυση συνεργασίας. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Έτος Τουρισμού Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνας. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ οργανισμών, μεταξύ περιφερειών, μεταξύ χωρών, ε, μεταξύ αυτών που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις, μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ο οργανισμός μας είναι έτοιμος να συνεργαστεί μαζί σας για να το πετύχουμε αυτό. Προσβλέπω λοιπόν την ενίσχυση της συνεργασίας μας που θα αρχίσει με το μνημόνιο κατανόησης που θα υπογραφεί αύριο στην επίσημη τελετή. Αυτό θα είναι όντω ένα επίσημο βήμα. Από την άλλη μεριά όμως βλέπω εδώ πολλά φιλικά πρόσωπα και ελπίζω να συνεχίσετε να μας στηρίζετε. Ήσασταν στη Γενική Συνέλευση και η φιλία σας και η στήριξή σας ελπίζω να συνεχιστεί για να κάνουμε πολλά ωραία πράγματα μαζί και να έχουμε καλά αποτελέσματα όπως είχαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να σας ξαναδώ αύριο και στη Μαδρίτη, στην έδρα μας. Να ξέρετε ότι είσαστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες σας. Διότι υπάρχουν πολλοί ε, κατάλληλα άτομα που ε, διευκολύνουν τη συνεργασία του Ευρωκοινοβουλίου ε, με τον ΠΟΕ και τον ΟΗΕ. Έχουμε και τον κύριο Ήμπρελ εδώ, ο οποίος είναι διευθυντής για το για τον κλάδο αυτό του ευρωπαϊκού τουρισμού. Ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να παρέμβουν. Κύριε Βάντεν Κάμπ, α, είπατε ότι θέλετε να μιλήσετε. Τι γκριμάτσα είναι αυτή. Ρωτήστε όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Είμαι πάντοτε πρόθυμος. Πάντοτε. Οι κυρίες προηγούνται. Η κυρία Ταπαρντέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο Κοινοβουλίο. Είναι προφανές ότι όταν μιλάμε για τουρισμό σήμερα θεωρούμε όλοι ότι είμαστε φίλοι και είμαστε μέλη στην ίδια ομάδα. Από την αρχή της ε, θητείας μου εδώ, η Κλάουντια, ο Ιστβαν, όλοι θελήσαμε να έχουμε μία ε, προσέγγιση συνολική, οργανωμένη. Ο τουρισμό δεν μπορεί να είναι τουρισμό των Αμερικάνων ή κάποια συγκεκριμένη χώρα. Πρέπει να είναι διεθνή, παγκόσμιο τουρισμό. Γι' αυτό είναι σημαντικό να καταρτήσουμε αυτόν τον διάλογο μεταξύ μόνο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εκπροσώπων τους και του δικού σας του οργανισμού στον κλάδο του τουρισμού. Είναι πολλά τα προβλήματα σήμερα στον τουρισμό προβλήματα που έχουν να κάνουν με νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας που ίσως ευνοούν ακριβώς την αλλαγή στις συνήθειες του τουρισμού. Στην Ευρώπη ανησυχούμε με πολλά εμπόδια, πολλές προκλήσεις, η τρομοκρατικές επιθέσεις λόγω χάρη, η ε, αίσθηση ότι δεν υπάρχει αρκετή ασφάλεια. Τα περασμένα χρόνια μπορέσαμε όλοι να διαπιστώσουμε ότι ο τουρισμός επιτρέπει τη δημιουργία δεσμών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ διαφορετικών υπήρων, δημιουργεί γέφυρες και διάβλους επικοινωνίας, αλλά και νέε τεχνολογίες, οι νέες μορφές τουρισμού δημιουργούν μια σειρά από προκλήσεις. Χαίρομαι πολύ που για σας η εκπαίδευση είναι μια προτεραιότητα. Ξέρετε ότι τα κράτη-μέλη μας θεωρούν ότι η κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού είναι προτεραιότητα. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν υπολογίζαμε και στοχεύαμε στην ε, ε, βελτίωση των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού, ιδίω για τους νέους που εργάζονται στον κλάδο αυτό. Υπάρχει και μια σχετική πρωτοβουλία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Τουρισμού και θα ήταν χρήσιμη η εμπειρογνωμοσύνη σας από τον ΟΗΕ για να μπορέσει να ευοδοθεί αυτό το εγχείρημα, διότι ο οργανισμός σας έχει πολύ σχετική πείρα. Θα είχα πάρα πολλά να πω, αλλά δεν θα τα πω. Αύριο θα υπογράψουμε ένα σχετικό μνημόνιο και αυτό θα είναι μια φάση επίσημη για να καταλήξουμε σε μια κοινή θεώρηση για τον ευρωπαϊκό και διεθνή τουρισμό. Γιατί όπως είπα δεν είναι καλό να μιλάμε για τουρισμό των Ευρωπαίων, τουρισμό των Αμερικανών, αλλά για τουρισμό γενικότερα. Ένα κλάδο ισχυρό στο διεθνές επίπεδο και όπου ούτως ή άλλως απασχολεί δεκάδες εκατομμύρια συμπολιτών μας σε αυτόν τον πλανήτη. Και ενδιαφέρει δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες που επιλέγουν ε, να ταξιδέψουν για να ψυχαγωγηθούν. Γι' αυτό θέλουμε ο τουρισμός να είναι και βιώσιμος. Πάρα πολλά θα είχα να πω, αλλά δεν θα τα πω. Και πάλι σας καλωσορίζω στην οικογένειά μας, είσαστε φίλος. Ευχαριστούμε, Κλάουντια. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μοντέιρο. Έχουμε δύο πολύ όμορφες και πολύ δυνατές προσωπικότητες που λέγονται και δύο κλάουδια στην Επιτροπή μας. Ναι. Αλλά με αυτές τις φιλοφρονήσεις από τον ε, ε, συνάδελφο Ιστβάν, όταν έχουμε τόσο εξαίρετους συναδέλφους γύρω μας, τα πράγματα περιπλέκονται. Καλώς ήρθατε λοιπόν ε, στο Κοινοβούλιο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το Γενικό Γραμματέα παγκοσμίω ενός κλάδου που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια της θητείας μας. Τον συζητάμε, ε, ορίζουμε προτεραιότητες, ε, την προσοχή, εφιστούμε την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους στόχου που θα πρέπει να εντοπίσει για την οικονομία των διαφόρων περιοχών και την τοπική οικονομία της Ένωσης. Βλέπω σήμερα ότι έχουμε παρόμοιες προτεραιότητες εμείς και εσείς στην διεξαγωγή των ύπατων ε, καθηκόντων σας. Θα πρέπει λοιπόν ε, θα μπορούσαμε λοιπόν να ε, συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας. Με όσα μας απαριθμίσατε, συμμερίζομαι και εγώ τον ενθουσιασμό σας και την ε, διάθεσή σας. Συζητάμε και εμείς εδώ αρκετά από τα βασικότερα θέματα και αναφέρθηκε η ασφάλεια, το θέμα των πολιτικών θεωρήσεων, η αρχή της αμοιβαιότητας, σε αυτό ακριβώς το έτος που μόλις ξεκίνησε για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας στον τουριστικό κλάδο και είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε σχέσεις και μορφές συνεργασίας μεταξύ λαών και τουριστών. Είναι σημαντικά θέματα αυτά για μας. Ακολουθούμε αυτή την συλλογιστική του βιώσιμου τουρισμού και τη μελετάμε. Να ενδιαφέρει πώς επίσης το θέμα των μεγάλων δεδομένων της ψηφιοποίησης μπορούν να απορροφηθούν σωστά από τον κλάδο. Θέλουμε καλύτερη συγκέντρωση πληροφοριών, στατιστικά δεδομένα, ώστε να μπορούμε στην Ευρώπη, με την ιδιαιτερότητα του κάθε για τους μέλους βεβαίως, να συνδυάσουμε τις πληροφορίες και να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες σε όσους έρχονται να μας επισκεφθούν. Επειδή είμαι από το ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα πρέπει να επισημάνω ότι για μας επίσημη προτεραιότητα είναι να υπάρχει μια ίδια γραμμή χρηματοδότησης για τον τουρισμό. Θέλουμε να δώσουμε την προσοχή που του αξίζει σε αυτόν τον κλάδο για να υπάρξει ακριβώς και ενίσχυση στο επίπεδο των κοντελίων. Πρέπει να υπάρχει μια πολιτική κοινή, κοινή ως προς κάποιους όρους, κάποιους στόχους του τουρισμού. Όμως αυτή η ενίσχυση του προπολογισμού, αυτή η δημοσιονομική ενίσχυση Ίσως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φωτίζεται από τη δική σας πείρα θα ήταν κάτι το πολύ χρήσιμο για να δούμε αυτή η δημοσιονομική ενίσχυση να είναι εύστοχη. Και εκ μέρους του ΕΛΚ να πω ότι εργαζόμαστε για το πώς μπορούμε να προασπιστούμε περισσότερο τον κλάδο και είμαστε διαρκώς πρόθυμοι με άλλους συναδέλφους και όλες τις πολιτικές δυνάμεις να υπερασπιζόμαστε τον κλάδο του τουρισμού, διότι είναι γνωστά τα ωφέλη του ως προς την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και τις μορφές συνεργασίας. Πολύ σας ευχαριστώ, αλλά έχουμε πέντε λεπτά ακόμη. Να δώσω το λόγο στον κύριο Πασκουάλ Τεγκράντες. Ή Πασκουάλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Το ερώτημά μου μπορεί να είναι κάπως ε, προκλητική. Κύριε Γενική Γραμματέα, νομίζω ότι είστε στην καλύτερη θέση να απαντήσετε, γιατί είστε σε ένα πολιτικό οργανισμό διεθνή, άρα η ΟΗΕ είναι ο καλύτερος για να απαντήσει. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Τουρισμού, Ευρωπαϊκής Ένωση ε, Κίνας. Ανοίγει τις πόρτες της επίσης η Κούβα στον κόσμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάθε προσπάθεια, όχι μόνο όμως, αλλά και είπα για να έχουμε μια νέα πολιτική κατάσταση στην Κούβα με καλύτερες προοπτικές και μεγαλύτερο άνοιγμα σε ό,τι αφορά τα τουριστικά ζητήματα. Χαιρόμαστε που έρχονται οι Κινέζοι στην Ευρώπη και του υποδεχόμαστε με ανοιχτέ αγκάλε. Όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο και μακάρι το ίδιο να γίνει και με του ε, Κουβανού, αν του αφήσουν βέβαια. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό μπορούμε και εσείς μπορείτε σε αυτές τις σημαντικές χώρες άλλες για πολιτικο-οικονομικό βάρος και άλλες για συμβολικούς λόγους, τόσο σημαντικές αυτές τις χώρες λοιπόν, πώς μπορούμε να επηρεάσουμε ώστε να κάνουν και οι Ευρωπαίοι ε, δουλειές στην Κίνα ή στην Κουβά. Να υπάρχει μια αμοιβαιότητα. Διότι πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα να έχει κανείς έναν εταίρο από την Κίνα ή από την Κούβα στην Ευρώπη. Θα έπρεπε λοιπόν σε αυτό το τομέα να ανοίξει κάπως ε, ε, ο δρόμος για την αμοιβαιότητα στις δημερισχέσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ντεγκράντες. Κύριε Γενική Γραμματέα, έχετε το λόγο. Τρία λεπτά έχουμε μόνο στη διάθεσή μας. Τρεις ήταν συμμετέχοντες και τρία τα λεπτά σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε τέτοιου είδους συναντήσεις ε, και πιο συχνά. Ίσως μία φορά το τρίμηνο ή το εξάμηνο είναι μια ιδέα που είχα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και ενδιαφέρον να συναντιόμαστε. Σε ό,τι αφορά την πρώτη Κλάουντια, φυσικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της ασφάλειας και η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο. Ήδη έχουμε το σχετικό ίδρυμα στην Ανδώρα και θα προσπαθήσουμε η δραστηριότητά του να επεκταθεί. Είναι ένα ίδρυμα που ασχολείται όμως με την εκπαίδευση και σίγουρα θα αξιοποιήσουμε την πλατφόρμα αυτή για να επεκταθούμε σε όλο τον κόσμο. Είχαμε στην Πορτογαλία μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση για πρώτη φορά ε, είχα ε, την επίσκεψη αυτή στη Πορτογαλία που τα πηγαίνει πολύ καλά και ένα από τα πρώτα εκπαιδευτικά κέντρα θα ανοίξει στο Εστορίλ. Το στηρίζει η πορτογαλική κυβέρνηση. Αυτό είναι ίσως ένα από τα πρώτα παραδείγματα για να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικά ισχυρά και ποιοτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Σε ό,τι αφορά τα big data, τα μεγάλα δεδομένα, δεν έχουμε δυστυχώς κάποιο τμήμα που να ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσουμε ξεκινώντα με αυτή τη νέα δομή που θα υποβάλουμε το Μάιο στο Εκτελεστικό Συμβούλιο ε, ένα ειδικό τμήμα. Με αυτό θα ξεκινήσουμε για την καινοτομία και την ψηφιοποίηση. Το ψηφιακό θεματολόγιο αν θέλετε για την οργάνωσή μα Κάτι νέο για εμά θα αυτό αλλά θέλουμε να κινηθούμε με γρήγορους ρυθμούς. Και νομίζω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον ε, κοινό και από τη δική σας πλευρά. Πολλές χώρες έχουν κάνει πολλά, έχουν κινηθεί προς αυτή την ε, κατεύθυνση και θα έχουμε άμεση συνεργασία μαζί τους. Για το δικό σας ερώτημα, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετές ευκαιρίες, στα ισπανικά ο και έχουμε και ζήτηση και από την Κούβα και από την Κίνα. Ιδίω για την Κούβα, ισπανικές ε, εταιρείε, αλλά ευρωπαϊκές γενικά. Το 80% των ευρωπαϊκών εταιρείων που δραστηριοποιούνται εκεί είναι ισπανικές. Και σίγουρα υπάρχει μεγάλη αλλαγή σε ό,τι αφορά το επίπεδο ποιότητας ε, των υπαρχόμενων υπηρεσιών στην Κούβα και συμφωνώ ε, με αυτό που είπατε. Απλά εμείς από τη δική μας θέση δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τέτοιου είδες σχέσεις. Αναλύουμε όμως τις μελλοντικές ε, δυνατότητες και ευκαιρίες για τον τουρισμό, που το μέλλον του σημαίνει επενδύσεις. Και γι' αυτό εξετάζουμε το δεχόμενο να καταρτήσουμε κοινά έργα και σχέδια με τις ε, αναπτυγμένες χώρες για την ανάπτυξη του τουρισμού σε αυτές τις περιοχές. Δεν υπάρχει ε, τέλος στον τουρισμό, είναι άπειρο το πεδίο και μπορούν οι διεθνείς επιχείρησεις να δραστηριοποιηθούν ε, παντού. Δεν ξέρω αν κατάλαβα πολύ καλά την ερώτηση που είχε να κάνει με την Κίνα και την Κούβα, αλλά εμείς θα είμαστε πολύ ενεργοί και θα προσεγγίσουμε ε, τις χώρες αυτές. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι με όλες τις χώρες μέλη. Να δούμε ποια αιτήματα έχουν. Να τις στηρίξουμε. Και όχι μόνο να αναλύσουμε, αλλά να παρέχουμε και την απαιτούμενη υποστήριξη στις χώρες. Επενδύσεις, περισσότερη τουριστική ποιότητα. Πολλά πράγματα αναλύουμε όλες τις δυνατότητες και όλες τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη του τουρισμού και των χωρών. Στα αγγλικά. Ξέχασα κάτι σημαντικό για το οποίο χρειαζόμαστε τη δική σας υποστήριξη. Χρειαζόμαστε περισσότερα ε, κράτη από την Ευρωπαϊκή και από την Ευρώπη. Αυτή είναι μια προσωπική παράκληση. Και κάτι άλλο που θα θέλαμε θα ήταν περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ε, να προσχωρήσουν στον οργανισμό μας, ε, ε, μεταξύ των νέων χωρών μελών. Τώρα για τη στρατηγική, για το πώς μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία και γέφυρες επαφής, αυτό θα το δούμε. Αλλά αν μπορείτε να μας υποστηρίξετε εσείς από εδώ θα ήταν κάτι πολύ θετικό. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γενική Γραμματέα. Ήταν η πρώτη συνάντηση για μας εδώ σε μια επίσημη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής ε, ΤΡΑΝ Μεταφορών και Τουρισμού. Ελπίζω να μην είναι τελευταία και να σανθούμε πολλές φορές και στο μέλλον. Αργότερα δεν θα έχουμε μετάφραση, θα τα πω αγγλικά. Ούγκρος, ορίστε. Η Κλάουντια Μοντέρο μίλησε για τη σημασία καλών μετρήσεων. Εδώ έχουμε ένα πολύ καλό ε, φυλάδιο που δημοσίευσε και η Κομισιόν, έχει υποστηρίξει για τις τάσεις τις τουριστικές ε, από το UNWTO. Εκδίδεται κάθε δεύτερο μήνα. Το έφερα ε, το τελευταίο τεύχος. Πέρυσι είχαμε έξι τεύχη και προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε όλο τον κόσμο και ιδίω στην Ευρώπη να ε, δώσουμε στοιχεία ώστε να μετρηθεί και να γίνει κατανοητό καλύτερα ο τουρισμός. Ευχαριστώ Ζόλταν, λέει ο Πρόεδρος. Μην ξεχνάτε ότι αύριο έχουμε μια ιστορική στιγμή στο Κοινοβούλιο και θέλω να σας ζητήσω να είστε μαζί μας με τον κύριο Ταγιάννη και τον κύριο Πολυκασβίλη στις 4. 4 το μεσημέρι. Αύριο. Ποια είναι η αίθουσα? 5B001. 5B001. Η ιστορική στιγμή, ε, η τελετή υπογραφής. Παρουσία του UNWTO. Ελπίζω να είστε και εσείς εκεί και θα τα ξαναπούμε στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Γεια σας.